monsieur le président de la république vous êtes Σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μας και μεγάλη ευχαρίστηση φυσικά που σας υποδεχόμεθα στην πόλη του Στρασβούργου. Χτες συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και η δική σας άφηξη λοιπόν εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης μας με την Αφρικανική Ένωση και φυσικά τις χώρες που την συνιστούν. Να υπογραμμίσω ότι έχετε κάνει εξαιρετική προσπάθεια στη χώρα σας. Βγήκατε από ένα εμφύλιο, ενισχύσατε τα όργανα της χώρας, το κράτος δικαίου, δώσατε δυναμική στην οικονομία, δημιουργήσατε μια βιομηχανική βάση, βελτιώσατε τους κοινωνικούς δείκτες. Η χώρα σας είναι μία από τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης στον κόσμο. 8% υπολογίζεται φέτος. Πρέπει να ε, είναι παράδειγμα για άλλες χώρες της Αφρικανικής Υπήρου και της Δυτικής Αφρικής. Βέβαια πολλά μένει να γίνουν. Η καταπολέμηση της φτώχειας, υποδομές, εκπαίδευση, υγεία, πρόσβαση στο πόσιμο νερό, και στον ηλεκτρισμό. Μην ξεχνάμε όμως ότι και η δική σας χώρα όπως και η Ευρώπη χτυπήθηκε από τρομοκρατικές επιθέσεις, ιδιαίτερα στον Γκραν Μπάσα. Πρόκειται για μια τεράστια μάστιγα, την οποία δεν θα μπορέσουμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό και μέσα από τις περιφερειακές οργανώσεις όπως η ε, Οργάνωση για τη Δυτική Αφρική ή η ίδια η Αφρικανική Ένωση. Η Ευρώπη και η Αφρική μοιράζονται τις ίδιες προκλήσεις σε πολλούς τομείς όπως το θέμα των μεταναστευτικών ροών. Θα πρέπει να δράσουμε στην ρίζα του προβλήματος, επενδύοντας περισσότερο και επενδύοντας καλύτερα στα πλαίσια μιας ουσιαστικής οικονομικής διπλωματίας για να δημιουργήσουμε ρυθμούς ανάπτυξης και απασχόληση. Η παρουσία της Προέδρου των Νίσον Μάρσαλ σήμερα το πρωί μας δείχνει τη σημασία που έχει η δράση μας για την αηφόρο ανάπτυξη και το κλίμα. Και η δική σας χώρα υφίσταται τις συνέπειες αυτές με ξηρασία, πλημμύρες και διάβρωση των παράκτιων περιοχών. Αυτά τα θέματα δημιουργούν προβλήματα στα δημογραφικά, στον τομέα της οικονομίας, της διαχείρισης των κρίσεων. Είναι τομείς τους οποίους θα εξετάσουμε στη συνάντηση κορυφής τον μήνα Σεπτέμβριο, Νοέμβριο μάλλον στο Αμπιτζόν στη συνάντηση κορυφής Ευρώπης-Αφρικής. Η παρουσία σας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι χαρά μας που είστε παρόν εδώ σήμερα. Να γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε ότι εμείς θέλουμε να βλέπουμε την Αφρική με αφρικανικό βλέμμα και όχι με ευρωπαϊκό βλέμμα. Γι' αυτό και η συνεργασία ανάμεσά μας είναι κρίσιμη και θα είναι κρίσιμη για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης και κατά των συνεπειών της κρίσης στον τομέα του κλίματος. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ Αντάνιο Ταγιάννη, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να απευθυνθώ στο σώμα σας, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεδριάζει σε Ολομέλεια. Είναι μια μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα και για τη χώρα μου να βρίσκομαι εδώ ενώπιον εκλεγμένων αντιπροσώπων πάνω από 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και αποτελείται εξαιτίας της πολιτιστικής σας ποικιλομορφίας, των πολιτικών σας δεσμεύσεων αλλά και της μεγάλης σας εμπειρίας ένα ιδιαίτερο ακροατήριο με υψηλό κύρος. Θέλω λοιπόν να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να σας μιλήσω για τις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Αφρική μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στη χώρα μου, την ακτή Ελεφαντοστού, η οποία έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως γνωρίζετε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, στι 25 Μαρτίου του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε στην αιώνια πόλη, τη Ρώμη, την 60η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Η συνθήκη αυτή σφράγισε την αλληλεγγύη μεταξύ των εθνών που μέχρι τότε βρισκόντουσαν σε πόλεμο. Οι ιδρυτές πατέρες λοιπόν της συνθήκης τη Ρώμη. η συνθηκη είχαν την ευφύ ιδρυτε πατερες λοιπον της συνθηκης τη ρωμη ειχαν την ευφυ ιδεα να βάλουν μαζί από κοινού τους πόρους, την ευφυΐα των ηγετών στην υπηρεσία της οικοδόμησης ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και ευημερία για όλους. Και η Ευρώπη αποτελεί πηγή έμπνευση για ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την Αφρικανική Ήπειρο. Δυστυχώς, τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τάση αναδίπλωση ταυτότητα σε πολλές περιοχές του κόσμου, είμαι πεπισμένο ότι εδώ, σε αυτό το ευγενέ σώμα, θα μπορέσετε να αντλήσετε την αναγκαία ενέργεια για να συνεχίσετε στο πνεύμα αλληλεγγύης, ανοίγματο και ειρήνης, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί σας. Αυτή η πεποίθηση βασίζεται στο γεγονός ότι από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπαψε να κοινωνεί στην ανθρωπότητα την πίστη της για έναν κόσμο ειρήνης, σταθερότητας και πρόδου. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απορμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012, αποτελεί μια αξιοσημείωτη απόδειξη γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, το μέλλον της ανθρωπότητας θα εξαρτηθεί από πολιτικές, από δράσεις και προγράμματα που μαζί θα καθορίσουμε στις χώρες μας, στις υπήρους μας, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Με άλλα λόγια, ο κόσμος θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε να γίνει. Γι' αυτό θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για τρεις μεγάλες προκλήσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον του πλανήτη μας και τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. εκεί μαζί σας αναφέρθηκε στα θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Οπότε δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω. Οι τρεις προκλήσεις για τις οποίες θα σας μιλήσω έχουν να κάνουν με την κλιματική υπερθέρμανση του πλανήτη, με τις μεταναστευτικές ροές και με την δημογραφική αύξηση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, πρώτη πρόκληση λοιπόν, η θέρμανση του κλίματος. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 Ηγέτε του κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι για να εγκρίνουν μια συμφωνία ιστορική σημασίας σχετικά με το κλίμα. Συμφωνία η οποία κυρώθηκε από μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών, μεταξύ των οποίων και ακτή του, η οποία ήδη έχει καταθέσει στον ΟΗΕ ε, τα της κύρωσης και η συμφωνία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία ιστορικής σημασίας για να περιοριστεί κλιματική αλλαγή. Σήμερα περισσότερο από ποτέ επίγει να υλοποιηθεί η συμφωνία αυτή, προκειμένου να περιοριστούν οι καταστροφικές συνέπειες της υπερθέρμανσης του κλίματος πάνω στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα. Η Ευρώπη πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή όταν επρόκειτο για παγκόσμιες προκλήσεις και τώρα μπορεί να δείξει το δρόμο. Η Ευρώπη μπορεί να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, την χρηματοδότηση, την τεχνολογία που χρειάζεται για την ενεργειακή μετάβαση προκειμένου να προχωρήσει ανεπιστρεπτή η συμφωνία αυτή του Παρισιού. Το Παρίσι μας έδωσε μια ιστορική σημασία σε ευκαιρία. Πρέπει λοιπόν να την υλοποιήσουμε. Σήμερα που σας μιλώ, βροχές, κατακλυσμοί πλήττουν τη χώρα μου και αποτελούν τη συνέπεια των κλιματικών αλλαγών. Οι καταστροφές είναι τεράστιες σε πολλές περιοχές της χώρας μου. Επίσης, πολλές περιοχές στην Αφρική αντιμετωπίζουν κύματα ξηρασίας που δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές για πολλές τοπικές κοινότητες που αναγκάζονται να μετατοπιστούν μαζικά. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, θέλω λοιπόν να σα ενθαρρύνω να συνεχίσετε να βάζετε το κλίμα στι προτεραιότητέ σα για να σταματήσει η τραγωδία αυτή που σήμερα παρατηρούμε ανά τον κόσμο. Πράγματι, υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να συνεχίσουμε σε έναν δρόμο προς μια πράσινη ανάπτυξη που χρησιμοποιεί ελάχιστο άνθρακα. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε περιορισμένα τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, χρησιμοποιώντας όμως και τους πόρους αυτούς για την οικονομική μας ανάπτυξη. Πρέπει μαζί να ενισχύσουμε την αντίσταση των κοινοτήτων μας, να μειώσουμε κάθε μορφή διακρίσεων, κυρίως σε βάρος των γυναικών. Πρέπει όλοι να φροντίσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές πιο αποτελεσματικής κατανομής και πιο ισόρροπες όσον αφορά τον πλούτο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, έρχομαι στη δεύτερη πρόκληση. Μια πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και είναι οι μεταναστευτικές ροές και η απασχόληση των νέων. Στη διάσκεψη της Βαλέτα για την μετανάστευση τον Εύρεο του 2015, εγώ είπα στους ε, επικεφαλείς που συμμετείχαν εκεί, τους μίλησα για δραματικά γεγονότα, για το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο ή στο ΣΑΕΛ, κάτι το οποίο απαιτεί περισσότερη αλληλεγγύη και συνεννόηση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική. Και γι' αυτό πρέπει να δράσουμε μακροπρόθεσμα και να αντιμετωπίσουμε όλους τους παράγοντες οι οποίοι προκαλούν αυτή την κατάσταση και γι' αυτό και επήγει να επανέλθει η ειρήνη και η ασφάλεια στην ε, ζώνη του Σαχέλ και της Σαχάρας και να ενθαρρύνουμε μία συνενετική πολιτική λύση στην σύγκρουση στη Λιβύη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι οι συγκρούσεις, το οργανωμένο έγκλημα δεν εξηγούν από μόνα τους τις μεταναστευτικές αυτές ροές που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια προς την Ευρώπη. Στους παράγοντες αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και τη φτώχεια, τη μιζέρια θα έλεγα, την ανεργία και το δημοκρατικό έλλειμμα που παρατηρείται σε πολλές χώρες. Και γι' αυτό την Δευτέρα 12 Ιουνίου του 2017 κατά την διάσκεψη τη, του G20 των 20 χωρών εταιρική σχέση με την Αφρική προτείναμε την δημιουργία ενός ειδικού σχεδίου που θα έχει σαν στόχο να διευκολύνει μαζικές επενδύσει υπέρ τη Αφρικής προκειμένου να δημιουργηθεί απασχόληση, κυρίως απασχόληση για τους νέους. Κάτι τέτοιο θα συνεισφέρει στη μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Δεδομένου λοιπόν της δέσμευσή της ε, για αυτό το σκοπό και επειδή ακριβώς μια τέτοια προοπτική είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλοί από εμά προτείναμε το σχέδιο αυτό να ονομαστεί σχέδιο Μέρκελ. Όμως διαπιστώσαμε ότι οι μεταναστευτικές ε, ε, ροές μέσα στην Αφρική είναι ακόμα μεγαλύτερες από αυτές που παρατηρούνται από την Αφρική προς την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η εκτήλεφαντος του υποδέχεται 5,5 εκατομμύρια ξένων στην επικράτειά της. Για 4 εκατομμύρια κατοίκους, που σημαίνει ότι είναι 26%. Η μεταφορά της διασποράς αυτής Αφρικανών έχει σαν αποτέλεσμα 1% του ΑΕΠ της χώρας. Όμως η αλληλεγγύη, η φιλοξενία της χώρας μου παραμένουν και έτσι βοηθούμε τις γείτονες χώρες. Η χώρα μου θα συνεχίσει να δείχνει αυτή την αλληλεγγύη απέναντι στους πληθυσμούς αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε στήριξη για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ε, θέσεις απασχόληση και να συνεχίσουμε να είμαστε μια χώρα φιλοξενίας και υποδοχής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η νεολαία αυτή η αφρικανική, η οποία ψάχνει την περιπέτεια στην Ευρώπη, συχνά αποτελεί το θύμα μαφιόζικων δικτύων και τρομοκρατικών οργανώσεων που τροφοδοτούνται ακριβώς από την ευάλωτη κατάστασή τους και την απογοήτευσή τους. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε απέναντι σε αυτούς τους νέους, να τους ενημερώσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν ότι είναι καλύτερα να παραμείνουν στην Αφρική από το να πάνε αλλού. Πρέπει επίσης να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 στο Παρίσι, στο Μέγαρο Σαγιό, που λέει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα μεταξύ τους μέσα σε εξωπρέπεια και σε κράτος δικαίου. Έχουν λογική και συνείδηση και πρέπει να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. Σε αυτό το πνεύμα ακριβώ ανοίγματο προς τη συνεργασία για πολλά θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος η χώρα μου θα σκίσει και την εντολή της το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την περίοδο 2018-2019. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλες τις χώρες σας για την μαζική στήριξη που προσφέρατε στην ακτή Ελεφαντοστού επί τη ευκαιρία της εκλογής μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η εντολή αυτή που αρχίζει την 1η Ιουνίου του 2018 θα τεθεί στον αστερισμό της ειρήνης που για τον λαό της ακτής του Ελεφαντοστού είναι η δεύτερη θρησκεία. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμοι Ευρωβουλευτέ, η τελευταία πρόκληση στην οποία θέλω να αναφερθώ είναι η δημογραφική αύξηση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις ε, του ΟΗΕ για το θέμα αυτό, ο παγκόσμιος πληθυσμός, ο οποίος σήμερα είναι περίπου 7,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, από τα οποία 1,2 δισεκατομμύρια είναι Αφρικανοί, θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια το 2056. Έτσι λοιπόν η Αφρική θα αντιμετωπίσει την πιο μεγάλη αύξηση που θα είναι 54% της δημογραφικής παγκόσμιας αύξησης μέχρι το 2050. Έτσι λοιπόν η αύξηση αυτή θα επιτρέψει στις μάλλον έτσι η Αφρική θα μπορέσει να φτάσει στα επίπεδα των πιο αναπτυγμένων περιοχών του κόσμου όπως είναι η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη. Η Νιγερία για παράδειγμα το 2050 θα είναι η πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό πριν από τη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδονησία και το Πακιστάν. Ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Αιθιοπία θα πάρουν τη θέση της Ρωσίας και του Μεξικού στον κατάλογο με τις 10 χώρες τις πολυπληθέστερες στον κόσμο. Για να καταλάβετε δηλαδή ποια θα είναι η θέση των τριών αυτών μεγάλων χωρών στην παγκόσμια κλίμακα μετά από λίγες δεκαετίες. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη λοιπόν θα είναι ακόμα πιο έντονη σχετικά με τους πληθυσμούς που είναι σε θέση να εργαστούν. Πράγματι ο ενεργός πληθυσμός στην Αφρική, την υποσαχαρική, θα περάσει από 5,18 εκατομμύρια σήμερα σε 1 δις 300 εκατομμύρια το 2050. Κυρίες και κύριοι, η Αφρική, κοιτίδα του πολιτισμού και της ανθρωπότητας θα παραμείνει η πιο νέα περιοχή του κόσμου μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Αυτή η διαπίστωση δημιουργεί προκλήσεις για όλους τους υπεύθυνους Αφρικανούς αλλά και για όλους τους πολιτικούς ηγέτες στον κόσμο. Η σταθερότητα της Αφρικής θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το θέμα της νεότητας της Αφρικής τις επόμενες δεκαετίες. Η δημογραφική ανάπτυξη δεν μπορεί να αγνοηθεί, πρέπει να συμπεριληφθεί στα προγράμματα ανάπτυξης και θα απαιτήσει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή την παιδεία, την ειρήνη και την επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει να γίνουν μαζικές επενδύσεις και στον τομέα των υποδομών, μεταξύ των οποίων ε, κάποια μεγάλα περιφερειακά σχέδια υποδομών στις μεταφορές, των εξηλεκτρισμό, την εκπαίδευση και την υγεία. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για την πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η χώρα μου, η οποία μετά από μια δεκαετία κρίσεων έχει βρει πια την ειρήνη. Έχει επίσης περάσει σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η πρόοδος αυτή είναι καρπός της κινητοποίησης των ίδιων των κατοίκων της χώρας. Η πρόοδος αυτή κατέστη εφικτή χάρη στην σημαντική τεχνική και οικονομική συνεισφορά των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της διακυβέρνησης, της γεωργίας και της ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω την δυνατότητα αυτή για να ευχαριστήσω όλος εγκαρδίως την Ένωση για την συνοδεία της όλο αυτό τον καιρό. Η εταιρική σχέση με την διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε στην χώρα μου να πετύχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, ο μέσος όρος ανάπτυξης της οικονομίας ήταν περίπου 9% ετήσια βάση και οι προβλέψεις για την περίοδο 2017-2020 βρίσκονται περίπου στο 7 8% το χρόνο. Ο πληθωρισμός έχει ελεγχθεί και είναι κάτω από 2% χάρη ακριβώς στην πρόσδεση στο ευρώ. Και ταυτόχρονα το έλλειμμα το δημοσιονομικό ελέγχεται περίπου στο 3% του ΑΕΠ. Φέτος η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική βέβαια, λόγω ακριβώς της χαμηλής, της πτώσης της τιμής του κακάου κατά 40% και είμαστε βασική παραγωγή αυτής της, αυτού του προϊόντος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε να ελέγξουμε τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Η χώρα μου είναι από τους πρώτους παραγωγούς στον κόσμο κάσουνατς και κακάο και θα γίνει επίσης και ε, ο πρώτος παραγωγός και για το ε, φινικέλαιο όπως επίσης και για το καουτσούκ. Είναι επίσης από τους καλύτερους ε, η χώρα μου στον τομέα των ε, βαθμολογήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είμαστε και σημαντικό hub παραγωγής ε, ηλεκτρισμού που θα περάσουμε από 2.000 ΜΒ το 2016 σε 4.000 ΜΒ το 2020. Έχουμε ένα από τα δίκτυα υποδομών τα πιο πυκνά και τα πιο ποικίλα στην Ευρώπη οδικά, λιμενικά, αερολιμενικά δίκτυα. Και έχουμε επίσης σημειώσει και σημαντική πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας, της, του αφοπλισμού των ατάκτων των παλαιών πολεμιστών. Ένα πρόγραμμα μάλιστα στο οποίο έχει συνεισφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν θέτουν σε αμφισβήτηση τις καλές ε, εξελίξεις. Ο δείκτης ασφάλειας της χώρας ε, είναι στο ίδιο επίπεδο με τη Γενέβη και τη Νέα Υόρκη. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συνεχιστούν και θα ενταθούν έτσι ώστε να υπάρξει μια δύναμη ασφάλειας ε, και τήρησης τάξης και στην χώρα μου. Κυρίες και κύριοι, λίγα χρόνια πριν από τη λήξη το 2020 της εταιρικής συμφωνίας του Κοτονού και τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να σκεφτούμε να υπάρξει μια νέα συμφωνία ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ορισμένες ιδέες οι οποίες εμπνέονται από τις υποδειγματικές σχέσεις που έχει η χώρα μου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχέσεις αυτές θα πρέπει να είναι ειλικρινείς, να εδράζονται στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη και φυσικά θα πρέπει κάθε χώρα να θέτει τους δικούς της στόχους. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν μέσα χρηματοδότησης ευέλικτα και να λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου και διαχείρισης που αν χρειαστεί θα πρέπει να ενισχύονται. Προφανώς εμείς θα έχουμε την δυνατότητα να εμβαθύνουμε τα θέματα αυτά αργότερα σε εύθετο χρόνο. Θα ήθελα πριν τελειώσω να προσκαλέσω όλες τις χώρες τις οποίες εκπροσωπείτε να πάρουν μέρος στην επόμενη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αφρικανικής Ένωσης τον μήνα Νοέμβριο στο Αμπιτζάν. Η σημαντική αυτή συνάντηση θα διεξαχθεί στα πλαίσια της παράδοσης φιλοξενίας της χώρας μου και θα είναι μια ευκαιρία αναφοράς και εξέτασης της διεθνούς συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας, ιδιαίτερα θέματα που άπτονται της νεότητας των χωρών μας και της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους παρόντες ε, ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ τον κύριο Ταγιάννη λοιπόν για την πρόσκληση την οποία μου απίθυνε. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτήν την εγκάρδια υποδοχή και από την σημαντικότητα της συμμετοχής σας εδώ παρουσία σας εδώ. Μου δώσατε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, όχι μόνο στην χώρα μου, αλλά και συνολικότερα στην Αφρικανική Ήπειρο. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον καθένα από σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ομιλία σας αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρωταγωνιστήσει στο διάλογο με τη χώρα σας και με την Αφρική. Σημεριζόμαστε τις προκλήσεις, ανεργία των νέων, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, παράνομης μετανάστευσης και κατά της κλιματικής αλλαγής. Υπογραμμίσατε τη σημασία που έχει επίσης η δημογραφική ανάπτυξη. Γι' αυτό και η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα στις δικές σας χώρες, αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα και να σας βοηθήσουμε να συνεργαστούμε για να μειωθεί η ανεργία στις χώρες σας και να δοθεί νέα ελπίδα σε όλους τους νέους Αφρικανούς το όνειρο των νέων Αφρικανών να μείνει στις χώρες τους δεν πρέπει να καταστραφεί εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Πρέπει να σταθούμε δίπλα σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξέρετε ότι θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι που ήρθατε. Να ξέρετε ότι έχετε εδώ φίλους και ότι η πόρτα μας θα είναι για σας πάντα ανοιχτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Α, υπάρχει ένα διαδικαστικό από την κυρία Φωνστόρ. Παρακαλώ, κυρία Φωνστόρ. Είναι διαδικαστικό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι στο άρθρο 31 του κανονισμού στο Προεδρείο τη Δευτέρα συζητήσετε μια έκθεση ότι το κτίριο του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες είναι σαφρό και θα, ενδεχομένως θα πρέπει να καταδαφιστεί. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Ε, δεν θέλω να πω ότι είμαι κατά της καταδάφησης του κτηρίου, αλλά θεωρώ ότι ως μέλη αυτού του σώματος πραγματικά έχουμε την αξίωση να δούμε και εμείς αυτή την έκθεση με